Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Καλημέρα σας καταρχήν. Εντάξει όλοι έχουμε πάρει τους καταλόγους ψηφοφορίας. Θέλετε λίγα λεπτά για να ετοιμαστείτε. Έχετε τις κάρτες ψηφοφορίας. Big news. Okay. Uh, so we have now to make Ας κάνουμε μια δοκιμή πρώτα. Αν έχετε έτοιμες τις κάρτες ψηφοφορίας, να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Can I... Okay, colleagues to vote. Okay, all group are... Ψήφισαν όλοι. Οι ομάδες εντάξει. Έγινε ο έλεγχο. Θα αλλάξουμε τη σειρά των σημείων. Πρώτα θα ψηφίσουμε το σχέδιο έκθεσης ε, του κυρίου Μορέλ για την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Βρήκατε τον κατάλογο ψηφοφορίας. Ξεκινάμε με την τροπολογία 41. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ τη 41 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ισοπαλία. Συμβαστική τροπολογία α. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Υπέρ, κατά. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε για καλό και για κακό. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται μάλλον. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 49. Άρχεται ψηφοφορία. Vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καλά που το ελέγξαμε. Τροπολογία 50. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά αποχές. Με την ίδια πλειοψηφία που νόμιζα ότι προηγουμένως ήταν πλειοψηφία, αλλά τελικά δεν ήταν από ό,τι φαίνεται. Δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμη. Τέλος ψηφοφορίας. Ισοπαλή, οπότε απορρίπτεται. Τροπολογία 52. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 11 άρχεται is ψηφοφορία Τέλος. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 20, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία closed. απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία Β. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Υπέρ της τροπολογίας 2. Στην άλλη σελίδα, γυρίστε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος της τροπολογίας 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Muy importante. <laughs> Gracias voting. You not I have to control ah. my colleagues. <laughs> is closed. Τέλος. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 31 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 33 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται με μία ψήφο πάλι διαφορά. 34. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Εγώ νόμιζα το έλκυ υπέρ. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για ή μάλλον σηκώστε πάλι τα χέρια για το 36. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η 36 εγκρίθηκε, τροπολογία 37. Ποιος είναι υπέρ. Ο έλεγχο έγινε για την 36 και τώρα ψηφίζουμε την 37. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά. Κατά τη γνώμη μου εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 39. Τέλος απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για τη 40, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται με 47 υπέρ, καμία αποχή και 8 νομίζω. Ε, κατά, ψηφίζουμε το νομοθετικό ψηφισμά, ψηφοφορία. η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, 51 υπέρ, κανείς κατά και δύο αποχές. Οπότε εγκρίνεται και συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία του κειμένου της προφορικής ερώτησης Εισαγωγή. Αρχικό κείμενο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρώτη ερώτηση. Το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ερώτηση 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και ερώτηση 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το κείμενο, όπως έχει τροποποιηθεί. Ηλεκτρονικά, έρχεται ψηφοφορία. Και ονομαστική ψηφοφορία, δεν κάνω λάθος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με 44 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 5 αποχές. Σχέδιο ψηφίσματος τώρα για την οριστικοποίηση της Βασιλείας Συμβαστική τροπολογία είναι ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία όμικρον υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία π, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Q σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας Q, άρχεται ψηφοφορία. Δεν χρειαζόταν καν ο έλεγχος. The oral amendment, sorry, I made a mistake. Α, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Είπα ότι ψηφίζουμε σε δύο τμήματα, ενώ έπρεπε να πω προφορική τροπολογία. Τώρα ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία. Καλώς με διορθώσατε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα, η συμβαστική τροπολογία χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε, με μεγάλη πλειοψηφία, η Πίτρο συμβαστική τροπολογία έχει εγκριθεί. Περνάμε στην 59. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία R, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία S, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία T, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 75, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία U, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία W προσθέθηκε ένα τέταρτο τμήμα. Θα το ψηφίσουμε και αυτό. Το πρώτο τμήμα Πρώτα, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, συγγνώμη. Επηρεάζεται και το πρώτο τμήμα από την προσθήκη, οπότε το πρώτο τμήμα χωρίς τη λέξη strong. Οπότε επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα χωρίς τη λέξη strong. Νομίζω ότι το τέταρτο το ψηφίσαμε μετά, αλλά επηρεάζονται όλα. Αλλά για τις τελευταίες στιγμής. Α, λάθος. Το πρώτο τμήμα δεν επηρεάζεται. Κάνω την προσθήκη, άρα δίκιο είχα. Το πρώτο τμήμα δεν έχει αλλάξει λοιπόν. Ποιο είναι υπέρ. Το είχαμε εγκρίνει. Άντε, επαναλαμβάνουμε κατά αποχής. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα τώρα. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα χωρί τη λέξη strong και μετά θα ψηφίσουμε ξεχωριστά τη λέξη strong. Δεύτερο τμήμα χωρί το strong. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα μόνο τη λέξη strong ω τρίτο τμήμα. Μόνο τη λέξη strong. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τέταρτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για το τέταρτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. This is the last sentence what we are voting now. Τελευταία πρόταση αυτή είναι που ψηφίζουμε τώρα για το CCF. Ψηφίσουμε μόνο τελευταία φράση, έτσι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στο συμβασμό Y. Η 91 αποσύρεται. Υπέρ του συμβασμού Y. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 95. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός Z υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβιβασμός AA σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά έχουμε το δεύτερο τμήμα με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείται με μία ψήφο παραπάνω. Τροπολογία 108 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Συμβασμός AB υπέρ κατά εποχές υιοθετείται. Τροπολογία 111 υπέρ κατά ελέγχουμε την 111. Μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Τροπολογία 112 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Το ΕΛΚ είναι υπέρ. Τότε το ελέγχουμε. Ελέγχουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία την 112. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Με μία ψήφο παραπάνω. Συμβασμός AC. υπέρ Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Παράγραφος 15. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Ψηφίζουμε τις αναφορές. 1 έως 9 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετούνται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά Ελέγχουμε την τροπολογία 1 ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Ο Σβέν πρέπει να είναι υπέρ, κανονικά. Πέρας ψηφοφορίες, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. 2 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 3 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. Αρχικό κείμενο Αναφορά 10 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Αναφορές από 11 έως 15 μαζί υπέρ κατά αποχές υιοθετούνται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Ουσιαστική νίκη και θα γιορτάσω μετά. Αναφορές από 16 έως 18 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετούνται. Τροπολογία 6. Αποσύρεται αυτή. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο. Αιτιολογική σκέψη A. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Αρχικό κείμενο, ε, αιτιολογική αναφορά B υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, συμβασμός C υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, συμβασμός D υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, συμβασμός E υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Προφορική τροπολογία EA της ΑΛΔΕ υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός F υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Συμβασμός G υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Τροπολογία 23 υπέρ, κατά, ελέγχουμε την 23. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 25. Ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Αιτιολογική σκέψη G υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείται. Συμβασμός I, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Συμβασμός J, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Συμβασμός K, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Τροπολογία 39, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Συμβασμός L, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Συμβασμός M, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Πέρας φοφορίας υιοθετείται. Δεν ψηφίσουμε τη 42. Πάμε να ψηφίσουμε το κείμενο με ονομαστική κλίση όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίσουμε τώρα. Πέρα ψηφοφορίας. 42 υπέρ, 5 κατά, 3 αποχές. Το ψήφισμα υιοθετείται. Και τώρα πάμε το σχέδιο νομοδότησης για τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για τη θέση του προγράμματο στήριξη διαφορετικών μεταρρυθμίσεων του Μαυρίδη. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ελέγχουμε την 27 με ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα. Vote closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Ένα, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε πέρας απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές δεκτή. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται να το επαληθεύσουμε τη ψηφοφορία. 166. Πέρας. Απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική π σε δύο, σι, σι, σε δύο μέρη υπέρ, πρώτο μέρος, κατά αποχές δεκτό, δεύτερο μέρος υπέρ, κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 186, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 187 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 188 υπέρ κατά αποχές δεκτή 189 υπέρ κατά αποχές δεκτή 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές δεκτή 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά 197 να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε πέρας απορρίπτεται συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ε σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Α, με συγχωρείτε, άρα η 50 έχει καταπέσει. Οπότε ψηφίζουμε κατευθείαν την 4. 4. Τροπολογία 4 υπέρ, υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε λοιπόν στο 54 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 55 υπέρ, κατά Δεν βλέπω την, ε, το EFTD, λοιπόν επαληθεύουμε την 55. Νομίζω απορρίπτεται, πέρας, απορρίπτεται, 56 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6, προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Νομίζω ότι την 59 δεν την ψηφίσαμε. Κατά τη γνώμη μου δεν ψηφίσαμε την τροπολογία 59. Is 59. Τροπολογία 59 κατέπεσε γιατί η 58 πέρασε γι' αυτό. Οπότε, μετά από την προφορική τροπολογία, στην τροπολογία 6, περνάμε κατευθείαν στην 77. Υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική G υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική H υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Την επαληθεύουμε. αρχή η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Μετά περνάμε κατευθείαν στην 94. Τροπολογία 94 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Πέρας απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, το ΕΛΚ είναι κατά. Να, ε, να την επαληθεύσουμε. Να επαληθεύσουμε την 95. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Άρα, μπερδεύομαι λίγο με τα χέρια. Απορρίπτεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Απορρίπτεται. 10 ε, και 102 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 αποσύρεται Πάμε λοιπόν στην ψηφοφορία του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 40 υπέρ 8 κατά μία αποχή συγχαρητήρια στον εισηγητή. Οπότε ολοκληρώσαμε τη συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίαση είναι Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 3 με 6.30 και τρίτη όλη μέρα. Σας ευχαριστώ. Λύεται τη συνεδρίαση.